Να συνεχίσουμε με τη σημερινή συνεδρίαση και περνάμε στο σημείο 10. Δέκτηση εφαρμογή σχετικά με την οδηγία του Συμβουλίου 2004-113 για την εφαρμογή τη αρχή τη μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίε και την παροχή αυτών. Η κυρία Κοσλόσκα είναι η συγκήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Το σημείο 6 δεν έχει συζητηθεί για τα θεμελιώδη δηλαδή δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το συζητήσαμε χθε. Uh, um, Μου λένε, λέει η Πρόεδρος, ότι αυτό το σημείο που έμεινε από εχθές θα το δούμε τελευταίο σήμερα. διότι σε αυτό το σημείο έχουμε εμπειρογνώμονες που είχαμε προσκαλέσει και επομένως πρέπει να μείνουμε στο πρόγραμμα. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε σχετικά με την έκθεση αυτή εφαρμογής της οποίας η συγγήτρια, όπω έλεγα, είναι η κυρία Κοσλόφσκα. Μιλάμε για μια πρώτη συζήτηση εν ώψη ενό εγγράφου εργασίας και ήθελα να δώσω την ε, δυνατότητα να γίνει μια πρώτη εισαγωγή στο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίε και κύριοι, η οδηγία αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες οδηγίες στην ε, νομοθεσία για τα, δικαιώμα... τα ίσα δικαιώματα. Ε, είναι μια οδηγία από το 2004, πάνω από 10 χρόνια δηλαδή. Και ήταν το πρώτο, η πρώτη νομοθεσία που ξέφυγε από την επαγγελματική ζωή και ε, περιέλαβε και άλλους ε, τομείς ισότητας ε, και ίσης μεταχείρισης ανδρών ε, και γυναικών. Αφορά τις υπηρεσίες οι οποίες δεν ρυθμίζονται από άλλα νομοθετήματα. Αφορά τις ε, ασφάλειες, συντάξεις, ιδιωτικά συνταξιδοτικά ταμεία, μεταφορές, παροχή υπηρεσιών, γενικότερα τον τομέα των μεταφορών, θυλασμό, μητρότητα, θέματα υγείας γενικότερα. υπηρεσίες στον χώρο του αθλητισμού, της διασκέδασης κτλ. Η οδηγία αυτή μπορεί όμως και να ισχύει για άλλους νέους τομείς οι οποίοι δεν υπήρχαν κατά την ε, περίοδο δημιουργίας της. Θα αναφερθώ συνοπτικά σε αυτούς, διότι στην έκθεσή μου θα χωρίσω τις υπηρεσίες σε τομείς, έτσι ώστε να μπορούμε να παρακολουθήσουμε καλύτερα τι συμβαίνει, ποιες είναι οι εξελίξεις σε κάθε τομέα. Και να δούμε την εξέλιξη της οδηγίας από την αρχή της μέχρι τώρα. Να δούμε τι πρόοδος έχει γίνει σχετικά με την εφαρμογή, τι χρειάζεται βελτίωση και πώς η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου ε, πρέπει να συνεχίσει. Και μετά θα περάσουμε στους νέους τομείς οι οποίοι δεν υπήρχαν κατά την ε, περίοδο ε, Δημιουργία τη ε, οδηγία. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Καταρχάς, πιστεύω ότι εδώ η οδηγία έχει μεγάλες δυνατότητες. Είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας εκείνος των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η οδηγία λοιπόν εδώ έχει επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα. Το άρθρο 5 της οδηγίας περιλαμβάνει στην αρχή του μία δυνατότητα παρέκκλησης. διαφορετική μεταχείριση ανδρών και γυναικών η οποία μπορεί να ισχύει σε ε, συγκεκριμένες περιπτώσεις, κατά εξαίρεση, όπως για παράδειγμα συντάξεις, ασφάλειες κτλ. Από το 2012, όταν η υπόθεση τεστ ΑΣΑ εκδικάστηκε υπήρχε πλήρης εφαρμογή του άρθρου αυτού και αυτό ήταν κάτι καινούριο, διότι εδώ πρόκειται για ασφάλιστρα στις ε, ασφάλειες υγείας, στα συνταξιοδοτικά ταμεία. Τα ασφάλιστρα αυτά για πολλά χρόνια ήταν διαφορετικά για άνδρες και γυναίκες ακριβώς εξαιτίας των διαφορετικών κινδύνων ε, υγείας και του διαφορετικού προσδόκιμου ζωή. Από το 2012 όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόσουν ε, παρόμοια νομοθεσία σχετικά με τα ασφάλιστρα, να ισχύουν τα ίδια ασφάλιστρα για άνδρες και γυναίκες. Αυτά μπορούν όμως να διαφοροποιηθούν βασισμένα σε άλλους παράγοντες κινδύνου για άντρες και γυναίκες. Όμως δεν μπορούν να είναι διαφορετικά εξ αρχής. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το καινούριο, κάτι το νέο στην, που επέφερε η οδηγία. Έπειτα, υπηρεσίες μεταφορών. Και όχι μόνο ε, την πρόσβαση, για παράδειγμα, σε δημόσιες συγκοινωνίες όταν κάποια γυναίκα έχει καροτσάκι με μωρό, αλλά και άλλα θέματα. Για παράδειγμα, ε, χώρους θυλασμού στις δημόσιες συγκοινωνίες, που μπορεί ε, να αλλάξει ένας γονιός πάνες στο παιδί του. Αυτές είναι οι συχνότερες και κυριότερες περιπτώσεις διακρίσεων κατά των γυναικών. Η σεξουαλική παρενόχληση είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, ιδιαίτερα στον χώρο των ε, μεταφορών. Και αυτό το θέμα μας έχει απασχολήσει αρκετά, ιδιαίτερα πρόσφατα, διότι υπάρχουν περιπτώσεις παρενόχλησης γυναικών σε τρένα, σε λεωφορεία, σε συγκοινωνίες. Η οδηγία λοιπόν θα εφαρμοστεί και εδώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θυλασμό και την προστασία της μητρότητας, εδώ νομίζω αξίζει να σημειωθεί ότι η οδηγία επεκτείνεται και σε άνδρες. Ωστόσο, θα ήταν καλό να αναφερθούν οι άνδρες συγκεκριμένα. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ε, μιλάμε για τους σταθμούς αλλαγής πάνας, αυ, τους χώρους αυτούς, αυτοί οι χώροι αναφέρονται μόνο ε, σε σχέση με τις γυναίκες. Δηλαδή, σε εστιατόρια, στις γυναικείες τουαλέτες υπάρχουν τέτοιοι χώροι αλλαγή πάνω Θα πρέπει να υπάρχουν και στις ανδρικές. Θα μπορούσαμε λοιπόν να εφαρμόσουμε την οδηγία και εδώ. Τώρα, ένας άλλος τεράστιος ε, τομέας είναι οι υπηρεσίες υγείας, οι οποίες καλύπτονται από την οδηγία. Και εδώ πρέπει να σταθούμε στην αναπαραγωγική υγεία και στις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται μόνο σε ένα φύλλο, ακριβώς εξαιτία της βιολογικής διαφοράς ανδρών και γυναικών. Από τη μία λοιπόν υπάρχει... υπάρχουν αμφιβολίες για το αν θα πρέπει να εφαρμοστεί η οδηγία σε αυτόν τον χώρο. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει Πολάκης ζητήσει να εφαρμοστεί η αρχή της επικουρικότητας στην αναπαραγωγική υγεία και ε, στο θέμα των αμβλώσεων. Από την άλλη όμως, η εγκυμοσύνη, ο θυλασμός, η προστασία της εγκυμοσύνης είναι κατηγορίες των υπηρεσιών υγείας που αφορούν μόνο γυναίκες. Προφανώς. Ωστόσο, η οδηγία αφορά και αυτούς τους τομείς. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω οι εμπειρογνώμονε μας να μας ενημερώσουν περισσότερο, ιδιαίτερα για το τι μπορεί να γίνει σε αυτούς τους ε, τομείς των υπηρεσιών υγείας που αφορούν αποκλειστικά γυναίκες. Και είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτό εγκαίρως έτσι ώστε να αποφύγουμε ε, περιττές συζητήσεις αργότερα που θα προκύψουν ακριβώς ε, από αυτή την οδηγία. Θα με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω λεπτομέρειες για την αναπαραγωγική υγεία συγκεκριμένα, διότι φοβάμαι ότι θα χάσουμε πολύ χρόνο για το θέμα αυτό. Εάν η οδηγία αυτή δεν εφαρμοστεί στην αναπαραγωγική υγεία, καλό είναι να μην ε, τη συζητήσουμε σε μεταγενέστερα στάδια εξέτασης της έκθεσης. Υπάρχουν τώρα ε, και άλλες υπηρεσίες. Ένας ε, κλάδος υπηρεσιών που αφορά την πρόσβαση σε γυμναστήρια, σε δισκοτέκ, σε μπαρ, σε σχολές χορού, όπου πολλές φορές οι τιμές εισόδου για άνδρες και γυναίκες διαφέρουν. Η οδηγία το επιτρέπει σε περίπτωση που αυτό βοηθά την συμμετοχή, την αύξηση της συμμετοχής ενός ή του άλλου φίλου. Γι' αυτό λοιπόν υποθέτω πως θα συζητήσουμε και αυτό το είδος υπηρεσιών. Όπως είπα και πριν, η οδηγία αυτή έχει τεράστιο δυναμικό και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για ορισμένους τομείς. Και πρέπει να πούμε ότι σε γενικές γραμμές εφαρμόστηκε σωστά η οδηγία. παρά το ότι υπήρξαν κάποια θέματα σχετικά με την εφαρμογή, όχι όμως ε, πολύ σημαντικά. Υπάρχουν ορισμένες ε, διατάξεις σχετικά με τις εθνικές αρμοδιότητες, όμως ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως όλη η οδηγία. Τώρα υπάρχουν κάποιες νέες υπηρεσίες για τις οποίες δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει, πώς θα εφαρμοστεί οι οδηγίες αυτές, οι ψηφιακές για παράδειγμα, Δηλαδή, τι γίνεται με τις διάφορες πλατφόρμες που επιτρέπουν επαφή μεταξύ των πελατών και των παρόχων υπηρεσιών. Αυτές οι υπηρεσίες βρίσκονται στα όρια της επαγγελματικής και μη επαγγελματικής ζωής, έτσι όπως προορίζει η οδηγία. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Airbnb. Τα νοικιαζόμενα δηλαδή διαμερίσματα, δωμάτια. Αυτή η πλατφόρμα βοηθά στην επικοινωνία ανάμεσα σε εκείνους που θέλουν να νοικιάσουν ε, το χώρο τους σε πελάτες. Μια άλλη περίπτωση είναι το Uber. Αυτές οι εταιρείες ε, διατείνονται πως είναι μια πλατφόρμα επικοινωνίας ανάμεσα ε, στον πάροχο και τον χρήστη της υπηρεσίας, ότι απλά βοηθούν στην επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστούν αυτές οι περιπτώσεις. Και είναι πολύ σημαντικό πιστεύω να το συζητήσουμε, διότι εάν η οδηγία καλύπτει και αυτές τις υπηρεσίες, τότε θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ισότητα των φύλων σε περισσότερους τομείς. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι με μεγάλη χαρά είδα πως οι προπαρασκευαστικές εργασίες έχουν εξελιχθεί με τόσο καλό ρυθμό. Όλοι όσοι συμμετείχαν έδωσαν πολύ σημαντικές πληροφορίες, συνεισέφεραν και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω την κυρία Καρατσόλο και όλα τα μέλη της ερευνητική μας ομάδας, καθώς και τους εμπειρογνώμονες. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Ευχαριστώ πολύ και την ε, Σιλβία Σπούρεκ από την Πολωνία, η οποία εκπροσωπεί και τον ε, διαμεσολαβητή για θέματα ισότητας φύλων. Ελπίζω να έχουμε μία διεξοδικότατη ε, επί της ουσίας συζήτηση, διότι θεωρώ πως αυτή η έκθεση θα αλλάξει πολλά προς το καλύτερο στην νομοθεσία σχετική με την ισότητα των φύλων. Έχει ήδη εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, σε έναν χώρο δηλαδή όπου πολύ συχνά παρατηρούσαμε διακρίσει ει βάρο των γυναικών. Και ελπίζω να αλλάξει την οπτική γωνία και την άποψη τη κοινωνία μα για την ισότητα των φίλων. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Καρατσόλο Ντιτορέλα από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ. Έχετε 10 έως 15 περίπου λεπτά για την παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Ε, χάρηκα ιδιαιτέρως που επεξεργάστηκα το θέμα αυτής της οδηγίας. Ε, θα ήθελα ε, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ως επιτοπλίστων συμφωνώ με όσα ακούσαμε μέχρι στιγμής και πιστεύω ότι είναι ε, είναι μια καμπή ε, αυτή η οδηγία είναι πελώριο το δυναμικό που έχει αναγνωρίζοντας ότι οι διακρίσεις μπορούν να ε, είναι και εκτός αγοράς εργασίας καλύπτουμε ε, ένα μέρος του χάσματος ανάμεσα στα δύο φύλλα. Ο, καθηγητής Μακόλγκαν χρησιμοποίησε αυτή την έκφραση το 2004, gap filling στα αγγλικά, ε, πλήρωση του κενού, του χάσματος ανάμεσα στα δύο φύλλα στα ελληνικά. Ε, δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, θα είμαι σύντομη. Είναι περιπετειώδες η ιστορία αυτής της οδηγίας. Σε πέντε χρόνια, αν θυμάμαι καλά, χρειάστηκαν για να συνταχθεί και... Στις αρχές του 2003 ήταν ευρύτερο το φάσμα των τομέων που καλύπτονταν Στο τελικό σχέδιο που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2004 προβλέπονταν διαφορετικοί τομείς ε, και με αυτό έπρεπε να συμμορφωθούν τα κράτη-μέλη. Ο στόχος είναι κατά πολέμηση της διάκρισης λόγω φύλου κατά την παροχή ε, αγαθών και υπηρεσιών και την πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες. Ε, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί βεβαίως, αναφερόμαστε στη συμβατική ε, ελευθερία και στην προστασία της προσωπικής και οικογενειακής ζωής και τις συναλλαγές που διεξάγονται στα πλαίσια της ελευθερίας της Αποκλείονται επίσης τα ΜΜΕ, η διαφήμιση και η παιδεία. Τα Ε και η διαφήμιση γιατί αποκλείονται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Αυτά τα αγαθά και οι υπηρεσίες διαφημίζονται στα μέσα ενημέρωσης και υπάρχει, υπάρχουν πολλές σεξιστικές ε, διαφημίσεις. Ε, θυμάμαι, δεν θέλω να κατονομάσω, αλλά μέσα υπήρχε μια πολύ μεγάλη διαφήμιση ένα αεροδρόμιο για μία οδοντόκρεμα. Οδοντόκρεμα και είχε γυμνές... <laughs> για ζυμαρικά. Ε, τι σχέση έχουν οι γυμνές γυναίκες με τα ζυμαρικά. Δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, ε, για την απασχόληση, για την ασφάλεια, για τις συντάξεις καλύπτονται αυτοί οι τομείς. Αναρωτιόμαστε, αφού καλύπτεται η απασχόληση, γιατί αποκλείεται η παιδεία. Υπάρχουν ε, εξαιρέσεις. Τι ξέρουμε μέχρι στιγμής. Το 2009 συντάχθηκε το τελικό σχέδιο, η τελική έκθεση. Ε, η πρώτη έκθεση για να γίνει η πρώτη αποτίμηση της κατάστασης για να μπορέσει να συνταχθεί το σχέδιο. Αυτά συνέβησαν πριν από μία δεκαετία. Μετά από αυτό έχουμε και άλλες εκθέσεις, αλλά με έμεση πληροφόρηση. Εκθέσεις ε, αναχώρα έχουμε το δίκτυο των ε, νομομαθών εμπειρογνώμων που μας ενημερώνουν, αλλά όχι ιδιαίτερα ειδικά για αυτή την οδηγία. Και είδα ότι για αυτή την οδηγία έχουμε μία-δύο σελίδες πληροφορίες μόνο. Άρα η τελευταία πλήρης έκθεση ήταν το 2009. Όχι μόνο επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος, αλλά επειδή έχει αλλάξει η κατάσταση, γι' αυτό ζητάμε στοιχεία. Τώρα ε, υπάρχουν διαφορετικού είδους υπηρεσίες που δεν υπήρχαν τότε. Και άρα δεν έχουν ε, συμπεριληφθεί, δεν έχουν ληφθεί υπόψη στην αρχική οδηγία. η εφαρμογή είναι copy-out, δηλαδή έχουν μεταφέρει ε, την ε, διατύπωση της οδηγίας ή έχουν ειδική νομοθεσία. Ποιο είναι το πρόβλημα ασαρφία. Ε, υπάρχουν δύο διαφορετικοί ορισμοί για τις υπηρεσίες, δεν υπάρχει ορισμός για τα αγαθά ή το αντίστροφο. Ε, κάποια κράτη-μέλη παρόλα αυτά και χαίρομαι γι' αυτό καλύπτουν ε, τα μέσα ενημέρωσης και την παιδεία στη δική τους εθνική νομοθεσία. Ένα άλλο θέμα είναι το gender reassignment, το περίφημο. Κάποια κράτη-μέλη ε, το συμπεριλαμβάνει στην νομοθεσία του, άλλα θεωρούν ότι καλύπτονται από την νομοθεσία για την ισότητα των δύο φίλων. Όμω δημιουργούνται προβλήματα. Δεν είχε καταγραφεί στην τράπεζα ένας τρανσεξουλ και άρα δεν είχε πρόσβαση ε, στις υπηρεσίες υγείας. Ε, ε, σεξουαλική παρενόχληση. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλοι συμφωνούν πως πρέπει η παρενόχληση να συμπεριλαμβάνεται. Όμως, όπως είπε και η συγγήτρια στο μετρό, στη, στο Λονδίνο, στο Παρίσι έχουμε πρόβλημα. Ποιος ε, φέρει την ευθύνη στον Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν πολλά πιλωτικά προγράμματα, το ξέρω για την αξιολόγηση, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει το θέμα κυρίως στη συνεργατική οικονομία, το, στο Uber παραδείγματος χάρη. Κοίηση και μητρότητα. Δυστυχώς δεν συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Ουσιαστικά ναι. Έχουμε προβλήματα ακόμη όμως. Στο Ηνωμένο Βασίλειο Έχουμε το Quality Act του 2010. Είναι η ειδική νομοθεσία. Απαγορεύονται οι διακρίσεις και παρενόχληση όταν θυλάζει η μητέρα. Ε, το δωματιάκι να αλλάξει την μπάνα. Το έχουν και στις αντρικές και στις ε, γυναικείες τουαλέτες. Και οι δύο μπορούν να επαναλλάξουν πάνω. Ε, προβλέπεται ειδικό χώρος. Όμως, όμως και το τονίζω, Πήγαινα στο δω, να πάρω το τρένο χθε. και είχα βάλει το ραδιόφωνο. Και έγινε μια φοβερή συζήτηση για κάτι που συνέβη το Σαββατοκυριακό. Θύλαζε μια γυναίκα στο Mother Care, είναι ένα μαγαζί με βρέφικα είδη. Και τη ζητήσα να πάει αλλού να θυλάζει. Δεν ξέρω αν τη ζητήσαν να πάει σε ένα ειδικό δωματιάκι, όμως ήταν πάρα πολύ ταραγμένη και ε, συγκλονισμένη. Είχα χρόνο και σταμάτησα το αυτοκίνητο γιατί με διέφερε τόσο πολύ η εκπομπή. Και πήγε ένας άντρα και είπε εγώ δεν θέλω να θυλάζει δίπλα μου στο εστιατόριο οποιαδήποτε γυναίκα. Δεν νιώθω άνετα. Ε, δεν, ε, μας, δεν υπάρχει σεβασμός. Μετά δυστυχώς δεν μπορώ να σου πω τι έγινε γιατί έκλεισα το ραδιόφωνο γιατί έπρεπε να μπω στο τρένο. Την ε, Κυριακάτικη εφημερίδα θα έχουν γράψει άρθρο, δεν το διάβασα. Τα λέω όλα αυτά γιατί. Γιατί ακόμη έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Για την κοίηση και για τη μητρότητα ήμουν συνεισηγήτρια για μία έκθεση και εκεί ε, ασχοληθήκαμε με το θέμα των αεροπλάνων. Ότι μετά από ένα ορισμένο αριθμό εβδομάδων δεν μπορούν να μπουν σε αεροπλάνο. Αλλά κυμαίνεται ο αριθμός των εβδομάδων ανάλογα με την αεροπορική. Δηλαδή μπορεί να έχετε ανταπόκριση και αν μπορείτε να μπείτε στο δεύτερο αεροπλάνο. time, so that Δεν έχουμε χρόνο όμως. Μήπως να τα πούμε αργότερα αυτά. Μου ζητήθηκε λοιπόν να εξετάσω τρία συγκεκριμένα ζητήματα, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, συντάξεις και συνεργατική οικονομία. Για το πρώτο και το τρίτο δεν είναι ξεκάθαρη απάντηση. Για το δεύτερο είναι σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Η υγεία είναι υπηρεσία. Η αναπαραγωγική υγεία όμως μπορεί να εκλειφθεί ως υπηρεσία. Και η εξωσωματική, αλλά και η άμβλωση είναι θέματα ε, αναπαραγωγικής υγείας. Είτε αποφασίζει κάποιος να μείνει έγκυος ή να ε, ξεγίνει και τα δύο υπηρεσίες είναι κράτη-μέλη όμως πρέπει να ρυθμίζουν κανονιστικά αυτές τις περιπτώσεις. Και γιατί, γιατί το λέω αυτό. Πριν από χρόνια ασχολήθηκα με αυτά τα ζητήματα και τρελάθηκα με τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Κάποια θεωρούν ότι είναι καθοριστικό για την ταυτότητα του ατόμου αυτό το ζήτημα. αλλά πάλι όχι. Αλλά, αλλά. Και το τονίζω γιατί είδα και τα στατιστικά στοιχεία. Στην Ευρώπη, ξέρετε, είναι φοβερός ο αριθμός των παιδιών που γεννιούνται παρένθετες μητέρες. Αν συνδυάσουμε δε και τις εξωσωματικές με τις παρένθετες, βλέπουμε πώς αυξάνεται ο αριθμός. Όμως στοιχεία δεν έχουμε ακριβώς ξεκάθαρα. Γιατί μπορεί να μην επιτρέπεται καν η παρενθετική. Τα βάζουν λοιπόν στο σακουλάκι της εξωσωματικής. Πού να βγάλεις άκρη. Για πηγαίνετε αλλού, για πήγε στην Ινδία, δεν είναι θέμα, θέματα αυτά. Πρέπει να ρυθμιστούν αυτά σε εθνικό επίπεδο. Ξεκάθαρη απάντηση δεν είναι. Δεν ξέρω αν μπορώ θετικά να σας πω, θα χρησιμοποιήσουμε την οδηγία. Μπορεί η διάκριση να ε, πάρει άλλη μορφή, αναπηρία, παραδείγματος χάρη. Αν δεν ε, έχει κάποια αναπηρία μια γυναίκα και δεν μπορεί να μείνει έγκυος και επι, ε, επιλέγει τη, μια παρένθετη μητέρα. Μήπως υπάγεται στην οδηγία για τις αναπηρίες. Όμως έχουμε και την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήταν πολύ στενή η ερμηνεία αυτού του ζητήματος. Δεν ήταν πολύ καλά τα νέα λοιπόν μετά την, αυτή, την απόφαση πρέπει τουλάχιστον περισσότερες πληροφορίες να έχουμε. Για πάμε στο δεύτερο σημείο σύνταξης. Άρθρο 5. Όπως είπε και η συγγύτρια, αυτή είναι η ουσία, αυτός είναι ο πυρήνας της οδηγίας, το ξέρουν όλοι αυτό. Με αυτή την οδηγία έχουμε τις αρχές στο άρθρο 5.1 και στο 5.2 είναι η εξαίρεση. Και τώρα μετά την απόφαση τέστασα, αποφάσισε το δικαστήριο να την βγάλει, να την αφαιρέσει από την εξαίρεση θετικό. Δεν είναι μόνο ασφάλειες, είναι γενικότερα χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ιδιωτικές, ε, ιδιωτικά συνταξιδοτικά ταμεία. Το 2004 είπαμε συντάχθηκε οδηγία και ισχύει για τα ιδιωτικά ταμεία. Μπορούμε να πούμε ότι αποκλείεται ως εκ τούτου επαγγελματική σύνταξη. Γιατί, γιατί υπάρχουν άλλες οδηγίες που καλύπτουν αυτό το ζήτημα. Όμως, Προς μεγάλη χαρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, διαπιστώθηκε ότι πολλά κράτη-μέλη χρησιμοποιούν αυτή την αρχή και για τις επαγγελματικές τάξεις. Ούτε εδώ είναι ξεκάθαρη η απάντηση. Πάμε στο τρίτο σημείο. Συνεργατική εικόνα. Φοβερό ζήτημα. Όλοι ξέρουμε τι είναι. Έχει φοβερά ωφέλη για τους παρόχους και για τους χρήστες. Πλατφόρμες στο διαδίκτυο και συναντιούνται οι πάροχοι με τους πελάτες. Uh, um, Uber και Airbnb συνεργατικές. Κατεβάζετε την εφαρμογή στο smartphone σας. Και τι κάνετε, μοιράζεστε το κόστος. Το Airbnb είναι για διακοπές, αν δεν το ξέρετε. Θέλετε να πάτε κάπου και θέλετε να ανταλλάξετε, θέλετε να βρείτε ένα δωμάτιο να μείνετε κάπου. για να πάτε στα ξένα. Τι γίνεται όμως με την παρενόχληση άμα γίνει μέσα στο αυτοκίνητο, πριν φτάσει εκεί. Ή δεν τη τον το δωμάτιο γιατί λέει δεν θέλω γυναίκες. Ή αντίστοιχα, αντίστροφα δεν θέλω άντρες στο δωμάτιό μου. Τι γίνεται τότε. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να ασχολείται και με αυτό το ζήτημα. Και έγραψε ένα πάρα πολύ καλό έγγραφο, αλλά Έχει μια σειρά σημείων εκεί, όχι όμως απαραίτητα και με το θέμα της ισότητας των δύο φύλων. δεν πρέπει να μας απασχολήσει και αυτό. Δεν πρέπει την ισότητα των δύο φίλων να την απασχολεί ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολλά τα ζητήματα που τίθενται. Έχω και μία διαφάνεια, προσπάθησα να αναλύσω την κατάσταση. Είναι εφαρμοστεί η οδηγία. Uber είναι υπηρεσία. Αν είναι υπηρεσία, τι γίνεται με την αποζημίωση, γιατί η υπηρεσία πρέπει να έχει οικονομική εμ, ανταμοιβή. όταν υπάρχει όταν μοιράζονται κάποιοι το κόστος για μια υπηρεσία, μπορεί να θεωρηθεί ως υπηρεσία. Εγώ νομίζω η απάντηση είναι διαφορετική. Πρέπει να δούμε τη σχέση της εταιρεία Uber με ε, τους παρόχους αφενός και τους χρήστες αφετέρου. Ναι, ένα, ένα, ένα λεπτό μόνο, δεν θα μακρηγορήσω. Airbnb τι είναι, είναι δημόσιο, ιδιωτικό, τι είναι το Airbnb. Και η σχέση πάλι είναι ανάμεσα στο Airbnb και τον πάροχο αφενός και το χρήστη από την άλλη. Μπορείτε να δείτε τις διαφάνειες. Μιλάω και για τις ε, ε, εξαιρέσεις. πολύ διαφορετικές ερμηνείες και άλλο πρόβλημα αυτό. Έχω δει και τις ε, ερμηνείες πολύ διαφορετικές. Άλλο πρόβλημα γι' αυτό. Θετική δράση, Πώς διβάξουν. Δεν έχουμε νομολογία δυστυχώς. Οι φορείς αρμόδιοι για την ισότητα των δύο φύλων έχουν καθοριστική σημασία. Ε, όμως δεν έχουν τον ίδιο ρόλο. Κάποιοι μπορούν να εκπροσωπήσουν πελάτες, κάποιοι όχι. Καλό θα ήταν να υπήρχε μια μεγαλύτερη ε, ομοιομορφία. Προτελευταία διαφάνεια. Ποιο είναι το συμπέρασμά μου. Αχ, συγγνώμη, είναι δύο διαφάνειες νωρίτερα. Ποια είναι τα συμπεράσματά μου. Συμφωνώ με την εισηγήτρια. δυνάμει φοβερή οδηγία. Αλλά πρέπει να το αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό. Και επίσης όχι μόνο στο χαρτί, να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία. Και πώς θα γίνει αυτό. Πλήρης τεκμηρίωση. Θέλουμε εκθέσεις να τεθούν τα ζητήματα όχι μόνο εφαρμόστηκε η οδηγία ναι ή όχι, πιο συγκεκριμένα στοιχεία, πώς εφαρμόστηκε, πού εφαρμόστηκε. Ξαναλέω, η οχι την ισότητα συγκεκριμενα στοιχεια να αντιβάσει εφαρμοστηκε Επιτροπή την ισότητα των δύο φύλων πρέπει να τη βάλει στους παράγοντες που εξετάζει τα πλαίσια τη συνεργατική οικονομία. Μόνο έτσι θα είναι επίσης όρις αυτή η οδηγία, όχι να θεωρείται ως παράρτημα στην νομοθεσία για το χώρο εργασίας, να ε, είναι εξίσου σημαντική. Τελευταία, τελευταία διαφάνεια, κάποιες πολύτιμε σκέψει μου. Μπορείτε να βαστείτε σε αυτή για να αναρωτηθείτε, να αναλογιστείτε τι γίνεται με αυτή την νομοθεσία. Την έχουμε, ωραία. Δίνουν πληροφορίες στα κράτη-μέλη. Τις ξέρουν πληροφορίες οι άνθρωποι που ασχολούνται με την οδηγία. Οι αρχές, τα μεμονωμένα άτομα, η νομολογία, η αποζημίωση, τι γίνεται. Είναι ικανοποιητική, είναι αποτρεπτική. Τελειώσω τώρα. Εκείνη η περίπτωση με το Mothercare, το μαγαζί. Ήταν εκεί και θύλαζε και της είπανε πηγαίνετε αλλού. Πολύ αμφιβάλλω αν ήξερε αυτή η γυναίκα που θύλαζε εκείνη την ώρα ότι ρυθμίζεται με τον νόμο αυτό που έκανε και ότι την προστατεύει ο νόμος. Ζητώ συγγνώμη. Έφαγα και πέντε λεπτά από τους υπόλοιπους. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος και θα δώσουμε την, τον λόγο στην κυρία Σπούρε και, και ακολούθως ε, θα έχουμε τις συνεισφορές από τα υπόλοιπα μέλη. Παρακαλώ. Uh, thank you very much. I'm really honored. Σας ευχαριστώ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που είμαι εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ε, πολλά λοιπόν ήδη ελέγχθησαν και ετέθησαν πολλά ερωτήματα Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι σύντομη. Έχω χωρίσει την παρουσίασή μου αφενός σε ένα τμήμα υλοποίησης και αφετέρου σε ένα τμήμα των σωμάτων των φορέων που είναι υπεύθυνα για την ισότητα και την ποιότητα και ένα τελικό τμήμα με κάποια συμπεράσματα και συστάσεις. Θα μιλήσω εξ ονόματος του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Πολωνίας και κάποιων άλλων φορέων ισότητας. Είμαστε μέλη του δικτύου Equinet, για το οποίο θα σας μιλήσω αργότερα περισσότερο. Εφαρμόσουμε λοιπόν την αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών για την ε, πρόσβαση και παροχή υπηρεσιών. Αυτά έχουν μετεγγραφεί από τα κράτη-μέλη, είτε υιοθετώντα νέα νομοθεσία, είτε τροποποιώντας υφιστάμενη νομοθεσία. Όμως αυτά αποτυπώνουν μόνο το υλικό πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και σε, ε, στην περίπτωση πολλών κρατών μελών ξεπερνά κατά πολύ το πεδίο εφαρμογή και τα ελάχιστα πρότυπα. Το 3-3 τη οδηγία λέγει ότι η οδηγία δεν θα εφαρμόζεται για το περιεχόμενο διαφημιστικό, μάλλον για διαφημιστικό περιεχόμενο, το οποίο κάθεται και από καλύπτεται και από την νομοθεσία κατά των διακρίσεων από την νομοθεσία χωρών όπως η Γαλλία ή η Ολλανδία. Κάποιες χώρες όπως η Ιρλανδία, η Λιθουανία και η Μάλτα καλύπτουν τις διακρίσεις αυτές και σε σχέση με τα μέσα επικοινωνίας. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν ενσωματώσει την, ε, το αποτέλεσμα της απόφασης τεστασά αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η μεταγραφή είναι απολύτω ικανοποιητική. Εγώ θα εστιαστώ στην προσέγγιση copy-out που ανέφερε και η προηγούμενη ομιλήτρια. Από Βέλγιο, Πολωνία, Ιταλία και Ρουμανία μεταξύ άλλων από τους εμπειρογνώμονες εκφράστηκε μια τοποθέτηση υπέρ της προσέγγισης copy-out που είναι μια αν θέλετε μινιμαλιστική προσέγγιση εφαρμογής. Ένα παράδειγμα τέτοιας ε, προσέγγισης είναι η πολωνική νομοθεσία. Η οδηγία εφαρμόστηκε το 2010 από την πράξη νόμου σχετικά με την εφαρμογή κάποιων από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ίση μεταχείριση. Είναι ο νόμος κατά των διακρίσεων ας πούμε. Υπό τον νόμο αυτό η ίση μεταχείριση επί τη βάση του φύλου της εθνικότητας ή του θρησκευτικού προσανατολισμού ε, συμπεριλαμβάνει τις υπηρεσίες και την πρόσβαση μεταξύ άλλων σε υπηρεσίες όπως η ενέργεια, οι διακρίσεις επί τη βάση αυτών απογορεύονται. Όμως, Απαγορεύονται επίση οι διακρίσει επί τη βάση αναπηρίας, ε, σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου κτλ. ηλικία για την πρόσβαση σε υγειονομικέ ε, και υπηρεσίες και υπηρεσίε παιδεία. Αλλά δεν απαγορεύονται οι διακρίσει ε, επί τη βάση των ίδιων παραγόντων όπως και πριν. σχετικά με το περιορισμένο πεδίο αυτού του, της πράξης νόμου κατά των διακρίσεων τοποθετήθηκε και το δικαστήριο. Συμπεριλαμβάνει η νομοθεσία αυτή ένα εξαρτητικό κατάλογο ε, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εφαρμοστεί ε, και όπως γνωρίζουμε όλοι οι ευρωϊκές οδηγίες δεν συνιστούν ένα πλήρες πλαίσιο προστασίας κατά διακρίσεων. Στην προσφυγή προς το συνταγματικό δικαστήριο λέμε ότι δεν θα πρέπει να καλύπτονται μόνο οι προϋποθέσεις συμμόρφωσης προς τις οδηγίες, αλλά και οι συνταγματικές διατάξεις. Στην Πολωνία τα πρότυπα προστασίας που προβλέπει το Σύνταγμα είναι υψηλότερα από τα πρότυπα που προβλέπουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Το Πολωνικό Σύνταγμα λέγει ότι δεν μπορεί να υπάρξει διάκριση κατά οποιοδήποτε σε στην πολιτική, κοινωνική ή οικονομική ζωή για οποιονδήποτε λόγο. Οι διατάξεις του... της πολωνικής νομοθεσίας σύμφωνα με την οδηγία που μεταφέρθηκε μπορεί λοιπόν υπό την έννοια αυτή να είναι αντισυνταγματικές. Και η πράξη νόμου με τις εξαιρέσεις και τα κενά που έχει θα μπορούσε να παραβιάζει και το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτή είναι η κίνδυνη λοιπόν μιας προσέγγισης copy-out. Οι φορείς ισότητος. Σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας όπως ξέρετε, τα κράτη-μέλη θα ορίσουν και θα προχωρήσουν σε απαραίτητες διαθετήσεις, απαραίτητες διαθετήσεις, σημαντική διατύπωση, σχετικά με, την, ε, με τους φορείς για την επιτήρηση, παρακολούθηση των, ε, της εφαρμογής των ε, κανόνων για την ίση μεταχείριση και για την αποτροπή των διακρίσεων. Χρειάζεται λοιπόν ανεξάρτητη βοήθεια αρρωγή προς τους ανθρώπους που υποβάλλουν καταγγελίες από τους φορείς αυτούς. Χρειάζεται διεξαγωγή ανεξάρτητων εκθέσεων και μελετών όπως και η δημοσίευση ανεξάρτητων μελετών και συστάσεων σχετικά με υφιστάμενα προβλήματα διακρίσεων. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την επαγγελματική εφαρμογή στο έδαφος χρειάζεται οι φορείς αυτή τη ισότητα να έχουν συγκεκριμένη εντολή και να είναι απολύτως ανεξάρτητοι. Η έλλειψη πόρων και προσωπικού εξακολουθεί να είναι ζήτημα σχετικά με την εντότητά του να προχωρούν σε έρευνα και έργο επικοινωνιακό στα θέματα αυτά. Η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της ε, για την EU Justice Agenda, το θεματολόγιο του 2020, περιγράφει το ρόλο που μπορούν να διαματίσουν οι φορείς αυτοί για τους πολίτες και η Κομισιόν θα συνεχίσει τη δουλειά της προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι φορείς αυτοί θα μπορούν να διαδραματίσουν το ρόλο αυτό μέσω της παρακολούθησης των ε, εφαρμοστείων ε, διατάξεων. Θα πρέπει επίσης να διαφημιστούν οι προϋποθέσεις και οι βασικές αρχές που θα διέπουν τα, τους φορείς αυτούς ισότητος και την ανεξαρτησία τους. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορέων αυτών έχει υπογραμμιστεί από τους ίδιους ως μια πολύ χρήσιμη πρακτική και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανταλλαγή των πληροφοριών και των βελτιστών πρακτικών, ε, δημιουργήθηκε το Equinet. Το δίκτυο φορών ισότητος, 45 συνολικά οργανισμοί από 33 χώρες με φορεί που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή συμμεταχείριση. Το 2012 και 2014 το Equinet προετοίμασε έκθεση για την εμπειρία των φορέων ή στην εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας, η στην εφαρμογη των διαταξεων τη οδηγια η μια εκθεση και η άλλη, για την στήριξη των παρόχων υπηρεσιών. Ποια ήταν λοιπόν τα συμπεράσματα και οι συστάσεις. Οι φορείς ισότητος χρειάζονται πρότυπα, πρότυπα αποτελεσματικότητας προκειμένου να εκπληρώνουν την εντολή τους. Η έλλειψη επαρκών πόρων είναι ένα πρόβλημα και χρειάζεται να διευρυνθεί, να υποστηριχθεί η δυνατότητα ε, ε, επιτήρησης και καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων οδηγίας. Υπάρχει και ένα θέμα ερμηνείας των διατάξεων της οδηγίας, γιατί δημιουργεί μια ασάφεια και σύγχυση μεταξύ των φορέων ισότητας. Επίσης υπάρχει έλλειψη ασφαλείας δικαίου σχετικά με τα υποκείμενα το διατάξεων της οδηγίας για την, ε, ως την ε, πρόσβαση και παροχή υπηρεσιών. Θα ήταν καλό σε όλα τα κράτη-μέλη ο ορισμός των αγαθών και υπηρεσιών να καλύπτει όλα τα σχετιζόμενα αγαθά και υπηρεσίε στον τομέα της υγείας και αυτά που χρηματοδοτούνται δημόσια και αυτά που χρηματοδοτούνται ιδιωτικά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ας πούμε. Στην Πολωνία είχαμε περιπτώσεις που αναφέρονται και στο ερευνητικό έγγραφο για γυναίκες που θύλαζαν δημοσία και που τους ζητήθηκε να βγουν από κάποιο εστιατόριο ή από κάποια άλλη δημόσια αίθουσα ανοιχτή στο κοινό. Πρέπει να καλύψουμε τέτοιες περιπτώσεις διακρίσεως και πρέπει να προχωρήσουμε σε μια ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την οδηγία αυτή, να προωθήσουμε το mainstreaming των φύλων προκειμένου να έχουμε περαιτέρω βελτιώσεις και διορθώσεις ε, στον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Και αυτό έχει σχέση με την αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας. Αλλά θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι οι εμπειρίες των φορέων αυτών δείχνουν την σημασία κάποιων περιοχών που δεν έχουν καλυφθεί ακόμα τα μέσα ε, τηλεπικοινωνιών, τη διαφήμιση και την παιδεία. Και θα ήθελα τέλος να υπογραμμίσω ότι κάποιοι φορείς υπογραμμίζουν ότι η ισότητα των φύλων είναι ένα ζήτημα που ακόμα δεν είναι απολύτως κατανοητό. Και η έλλειψη της ισότητας των φύλων είναι κάτι που δεν αναγνωρίζεται ευρέως ακόμα. Ελπίζω η έκθεση αυτή, οι απόψει αυτέ να είναι χρήσιμε για τη δουλειά σα και είμαι έτοιμη να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση θα μπορούσατε να έχετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τις δύο μιλήτριες για την ε, συνεισφορά τους. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στους σκιώδεις των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Ρίκνερ, αρχικά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τι ακριβώς κάνετε. Και πολλές φορές όταν ε, ακούμε με μεγάλη προσοχή μας δημιουργούνται και ερωτήματα. Και έχω και εγώ πολλά ερωτήματα. Πιστεύω πως για την Επιτροπή μας είναι ιδιαίτερα ε, ευχάριστο που πρόκειται για μια οδηγία η οποία στόχο έχει την ισότητα ανδρών και γυναικών. Και πρέπει να είμαστε στη θέση να δούμε τα αποτελέσματα στην πράξη της οδηγίας αυτής στους διάφορους τομείς, στους τομείς ε, των ε, υπηρεσιών. Βλέπω ότι η οδηγία αυτή στέφθηκε με επιτυχία. Όμως ο δρόμος ήταν δύσκολος. Έπρεπε να αναγνωρίσουμε τι ακριβώς είναι αυτή η ίση πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες και ε, κατά τη διάρκεια της ε, διαδικασίας συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες τις οποίες δεν μπορούσαμε να είχαμε προβλέψει λύνουμε το ένα πρόβλημα, προκύπτει το επόμενο. Είναι λοιπόν μια διαδικασία εν εξελίξει ακόμα η εφαρμογή της οδηγίας. Αναφέρατε κάποια παραδείγματα θετικών μέτρων, τα οποία θεωρώ πολύ σωστά. Αναφέρατε, νομίζω η πρώτη ομιλήτρια, ότι δεν υπάρχει αρκετό υλικό το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να συγκρίνουμε τις ε, περιπτώσεις εφαρμογής στα κρατημέλη. Οι γυναίκες σε, στο λέω Πολιτστάτ μπορούν να αγοράσουν εισιτήρια για ποδοσφαιρικούς αγώνες σε χαμηλότερη τιμή από ό,τι οι άντρες και η αιτιολογία ήταν ότι οι φύλαθλοι θέλουν περισσότερες γυναίκες, θέλουν να δώσουν κίνητρα στις γυναίκες για να παρακολουθούν τους αγώνες. Και από αυτήν την ε, πρωτοβουλία άλλαξε το φιλαθλοκοινό στους αγώνες στο Λεοπολτστάτ. Υπάρχουν λοιπόν τέτοια παραδείγματα θετικών μέτρων τα οποία οδηγούν στην επίτευξη του στόχου, δηλαδή στην μεγαλύτερη ισότητα ανδρών και γυναικών. Δεν πρέπει λοιπόν να έχουμε μόνο τον τελικό στόχο κατά νου, αλλά να δούμε και πώς μπορούμε με διάφορα μονοπάτια να φτάσουμε σε αυτόν. Να αλλάξουμε τις λεπτομέρειες και πιστεύω πως η σύγκριση με τα παραδείγματα διαφόρων χωρών, μικρά παραδείγματα, μπορεί να μας ανοίξει τα μάτια για να δούμε σε ποιες περιπτώσεις διαπιστώνονται διακρίσεις και πώς μπορούμε να τις ξεπεράσουμε, ποια είναι τα θετικά παραδείγματα. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι ίσως θα ήταν καλό να σταθούμε στην ε, περίπτωση των πολλαπλών διακρίσεων και να δούμε και εδώ ορισμένα θετικά παραδείγματα, παραδείγματα προς μίμηση. Ε, μπορούμε να εξετάσουμε το θέμα, για παράδειγμα, της μετανάστευσης των γυναικών προσφύγων. Πώς ε, εδώ υπάρχουν θετικές ε, πρακτικές. Να δούμε δηλαδή τις διαφορές. Φυσικά πρέπει να προσέχουμε τις, ε, πρέπει να προσέχουμε να μην δημιουργούνται ανισότητες ακριβώς λόγω αυτής της Θετική διάκριση. Τώρα, συνεργατική οικονομία. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Η οδηγία όταν ψηφίστηκε δεν είχε ιδέα το τι μπορεί να σημαίνει αυτή η συνεργατική οικονομία. Δεν υπήρχε ακόμα και οι νομικές συνέπειες ιδιαίτερα ως προς την ευθύνη δεν ήταν ακόμα σαφείς. Τώρα, εάν θα πρέπει να ε, Τώρα μάλλον θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις πλατφόρμες και να δούμε εάν σε περιπτώσεις όπως το Airbnb χρειάζεται ε, μια ε, πολιτική μηδαμινής ενοχής στις διακρίσεις. Τώρα, ο τομέα των υπηρεσιών υγεία είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι πρόκειται για ε, τομέα όπου κινούνται πολλά χρήματα. Τα φάρμακα είναι επίση ένα αρκετά επικερδή τομέα και πάρα πολύ σημαντικό. Και να δούμε πώς εδώ μπορούμε να ε, χρησιμοποιήσουμε τα θετικά μέτρα ως παράδειγμα. Επίσης, θυμάμαι ότι όταν είχε ψηφιστεί η οδηγία, μας έλεγαν ότι στον ασφαλιστικό τομέα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, διότι αναλογιστικά δεν μας βγαίνουν τα νούμερα και πρέπει να δούμε πώς ε, θα ε, γίνει. Και είναι πολύ δύσκολο. Ευτυχώς όμως δόθηκε λύση σε αυτό. Και όπως μας είπατε ότι στα κράτη-μέλη αντέδρασε ο νομοθέτης και ανέλαβε δράση. Εδώ βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει πως δεν θα πρέπει να έχουν οικονομικές επιπτώσεις. Δεν θα πρέπει η εφαρμογή της οδηγίας να έχει οικονομικές επιπτώσεις δυσάρεστες, να αυξηθεί το κόστος. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε πάντως και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ κυρία Σότροβα λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη μελέτη, για τα συμπεράσματα και για τις παρουσιάσεις. Εδώ έχουμε λοιπόν μια σειρά από διατάξεις, από ε, διατάξεις νομοθεσίας και θα πρέπει να δούμε τι αντίκτυπο έχουν όλα αυτά και η εφαρμογή τους. Νομίζω ότι η συγκήτρια προς την κατεύθυνση αυτή θα κινηθεί και επομένως ε, το έγγραφο θα, είναι, θα, ε, θα ενέχει τελικά μια προστιθέμενη αξία για την όλη δουλειά που γίνεται στο Κοινοβούλιο. Για την ε, υγεία τη σεξουαλική και αναπαραγωγική. σε αυτόν τον τομέα μιλούμε για όρους, εξετάζουμε δηλαδή έννοιες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών Υπάρχει ένα πλαίσιο κατά των διακρίσεων ευρωπαϊκό, αλλά εδώ έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα κράτη-μέλη. Η μελέτη μας λέει ότι έχουμε σημαντική αύξηση ε, του φαινομένου της χρησιμοποίησης των παρένθετων μητέρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει ότι αλλάζουν, ε, αλλάζει το ύφος, το στυλ της ζωής, αλλάζουν οι συνήθειες των ανθρώπων. Αλλά καλό θα ήταν να μην συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το παιδί είναι ένα αντικείμενο και έχουν το δικαίωμα να το έχουν ή να μην το έχουν και εν πάση περιπτώσει είναι κτήμα τους των γονέων δηλαδή δεν είναι ένα αγαθό δεν μπορεί το παιδί να το εξετάζουμε όπως ένα από τα υπόλοιπα αγαθά που εξετάζουμε στο πλαίσιο της πρόσβασης στην αγορά και της παροχής αγαθών και υπηρεσιών. Νομίζω ότι εδώ χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση φιλοσοφικά και δεν θα επιθυμούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί προς μια τέτοια κατεύθυνση. Νομίζω λοιπόν ότι στα πλαίσια της εξήτησης αυτής της οδηγίας καλό θα έπρεπε να μην ε, εξετάσουμε το θέμα υπό την οπτική αυτή. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου η άποψη. Ε, ε, πρόκειται για ένα πρόβλημα και επιστημονικό αν θέλετε και ιατρικό αλλά και ηθικό. Δεν πρέπει αυτό να είναι αντικείμενο λοιπόν μιας πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτό θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Ε, θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε κάτι άλλο ακόμα. Στο οποίο αναφέρθηκε η συγκέντρια ε, ή μάλλον η εμπειρογνώμων σχετικά με ένα κρούσμα ε, μητέρας που θύλαζε σύμφωνα με την νομοθεσία δεν μπορεί να απομακρύνεται από δημόσιο χώρο μια τέτοια μητέρα, μια μητέρα που θυλάζει. Ε, είναι μάλλον ίσως να μην υπάρχει νομοθεσία αλλά ίσως να είναι δυστυχές και ατυχές το οποίο δεν το προβλέπει η νομοθεσία. Εγώ η ίδια ε, τις φορές που χρειάστηκε να θυλάσω ε, απομακρύνθηκα από τους δημόσιους χώρους για προσωπικούς λόγους αν θέλετε γιατί δεν αισθανόμουν άνετα. Από εκεί και πέρα όμως η ελευθερία πρέπει να παρέχεται συνολικά. Δηλαδή η μία μητέρα θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να θυλάσει όπου επιθυμεί. Αλλά ίσως από την άλλη μεριά κάποιος θα μπορούσε και να ενοχληθεί. Θα έπρεπε λοιπόν στους κινηματογράφους, στα εστιατόρια, στους δημόσιους χώρους να υπάρχει πρόβλεψη μιας αίθουσα ενός δωματίου, ώστε το οποίο η μητέρα να είναι προστατευμένη και ήσυχη, ώστε αυτό να μην ενοχλεί οποιονδήποτε ούτε προς τη μία κατεύθυνση, ούτε προς την άλλη κατεύθυνση. Αλλά στο κέντρο της νομοθεσίας και της προστασίας πρέπει να είναι το παιδί, το οποίο εκείνο είναι που υπάρχει απόλυτη ανάγκη να θυλάσει. Πρόκειται όμως για ένα τόσο φυσιολογικό θέμα, ένα τόσο φυσικό θέμα, που θα έπρεπε να έχουμε μια προσέγγιση περισσότερο ανθρώπινη και λιγότερο νομοτεχνική, αν θέλετε. Είναι, θα ήταν ε, αρκετά θλιβερό να προβλέψουμε κυρώσεις, δηλαδή βάσει της νομοθεσίας για κρούσματα τέτοιου είδους. Δηλαδή αν φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο ίσως ε, εκφράζοντας, επαναλαμβάνω, μια προσωπική ανθρώπινη θέση ε, θα το έβρισκα κάπως ε, απόκληση στον ανθρώπινο τομέα. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, παρακαλώ να περιοριστείτε στο χρόνο που έχει προβλεφθεί, γιατί έχουμε και άλλη συζήτηση και δεν θα έχουμε χρόνο τελικά. Σας παρακαλώ ε, ξέρω ότι πάντα στο τελευταίο σημαίνει αυτό, να είστε λίγο πιο σύντομοι και πιο συγκεκριμένοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαστε και ο εισηγήτρια εδώ. Η συνάδελφός μου είναι και την αντικαθιστώ. Γι' αυτό λοιπόν ε, ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της. Η συνάδελφος και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, παρουσίαση αυτή, για την αναφορά σε όλες τις πτυχές της ε, οδηγίας σχετικά με την ε, παροχή υπηρεσιών. Είναι μια μεγάλη συζήτηση που συνδέεται με πολλά, με την συμφωνία για το ελεύθερο εμπόριο κτλ. Εγώ έχω δύο πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις για παραδείγματα. Η κυρία Ρέγνερ μας είπε ένα θετικό παράδειγμα από την Αυστρία, για παράδειγμα, με την διαφορά των τιμών στα γήπεδα. Είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά δύσκολο θέμα. Αυτή η διαφορά των τιμών, για παράδειγμα, δεν είναι όμως μόνο εκεί, είναι και στα κομμωτήρια. Και εδώ υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα. Όταν μια γυναίκα πάει για κούρεμα στην Αυστρία, το έχω δει και σε άλλες χώρες, ε, θα πληρώσει περισσότερα από ότι ένας άνδρας. Ακριβώς επειδή είναι γυναίκα, μόνο και μόνο λόγω του φίλου της. Μια γυναίκα λοιπόν ε, ε, με κοντά μαλλιά όταν πηγαίνει στο κομμωτήριο στην Αυστρία πληρώνει για κούρεμα περισσότερα από ότι ένας άνδρας με μακριά μαλλιά. Έχει προσπαθήσει το ε, εμπορικό επιμελητήριο να ε, παρέμβει, έχει χαρακτηρίσει την πρακτική ως ε, άδικη, όμως αυτή η οδηγία πιστεύω πως δεν καλύπτει αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν σε μένα προκύπτει το ερώτημα τι κάνουμε. Έχω δει και σε άλλες χώρες παραδείγματα στις τιμές, τιμές της αγοράς marketing δηλαδή. Όταν για παράδειγμα ένα προϊόν, δηλαδή ξυριστική μηχανή, αποσμητικό, ε, διατίθεται στην αγορά έχει διαφορετική τιμή για τις γυναίκες και όχι για, τις, ε, και για τους άντρες. Δηλαδή ένα αποσμητικό που ε, απευθύνεται σε γυναίκες είναι πιο ακριβό από ότι ένα αποσμητικό που απευθύνεται στους άντρες. Ελπίζω λοιπόν με αυτήν την οδηγία να μπορούν να προστατευτούν οι καταναλωτές ε, από αυτές τις διακρίσεις. Ε, σας ευχαριστώ κύριος Γκέρικ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση σήμερα και θα ήθελα να σταθώ στο δικαίωμα του θυλασμού. Αυτό που μας είπατε για την περίπτωση της Πολωνίας είναι κάτι που το γνωρίζω ως ευρωβουλευτής του οικογενειακού κόμματος και από τη Γερμανία, από την χώρα μου. Οι γυναίκες που θυλάζουν αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα όταν θέλουν να θυλάσουν δημόσια. Τις διώχνουν σε σιδηροδρομικούς σταθμούς. Έχουμε δει πολλές φορές ότι στέλνουν τις γυναίκες με μωρά στις τουαλέτες για να θυλάσουν τα παιδιά τους. Υπάρχουν προβλήματα λοιπόν τα οποία θεωρώ πως πρέπει να ε, επιληθούν. Ε, πριν από κάποιους μήνες, μαζί με κάποιους συναδέλφους, ε, συγκέντρωσα υπογραφές για τον θυλασμό, για τον ελεύθερο θυλασμό στην Ευρώπη. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να συγκεντρώσουμε αρκετές υπογραφές για να προχωρήσουμε, αλλά υπάρχει μία σφραγίδα ένα σήμα ε, που το βλέπετε εδώ για το δικαίωμα των γυναικών στον ε, δημόσιο θυλασμό. Είναι ένα αυτοκόλλητο ε, που σας δείχνω, το οποίο μπορεί κάποιος να κολλήσει στην πόρτα του ή σε κάποιο δημόσιο χώρο και με αυτό σηματοδοτεί ότι εδώ είναι ένας χώρος όπου μπορεί μια γυναίκα να θυλάσει το μωρό της. έτσι ώστε οι θυλάζουσες μητέρες να έχουν ένα καταφύγιο ώστε να μπορούν να θυλάσουν. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα, ε, μια ευρωπαϊκή νομοθεσία για το θυλασμό και η Μεγάλη Βρετανία μας δείχνει το σωστό δρόμο με ε, την, το Accessibility Act όπως λέγεται όπου ε, οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα στο θυλασμό και απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση. Πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε και στην Ευρώπη ένα, accessibility act, ε, μια νομοθεσία σχετικά με την πρόσβαση αυτή των γυναικών. Η ε, Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων πιστεύω πως πρέπει να αναλάβει το θέμα αυτό γιατί οι θυλάζουσες μητέρες χρειάζονται υποστήριξη, τη δική μας υποστήριξη. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να υποβάλουμε μια νομοθετική πρόταση από αυτού. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρου της Κομισιόν η κυρία Μαλέτρας. Oui, bonjour. Merci beaucoup de... Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Η Κομισιόν πολύ είναι ικανοποιημένη σχετικά με την με δουλειά του Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της ΟΔΙΑΓΕΣ αυτής 2413 όπως και της δημοσίευσης ε, του, από πλευράς του Κοινοβουλίου αυτής της μελέτης. Θα θέλαμε να διαφημίσουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει μέτρα για να μετεγγράψουν την οδηγία στην εθνική νομοθεσία και να προβλέψουν οργανισμούς και φορείς σχετικά με την εφαρμογή της. Εκτιμούμε ότι δεν είναι απαραίτητο να προταθούν αυτή τη στιγμή τροποποιήσεις ή τροπολογίες της οδηγίας, όμως χρειάζονται κάποιες διευθυνήσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τις εξαιρέσεις από την ε, αρχή ίσης ε, ε, μεταχείριση ανδρών και γυναιτών για την πρόσβαση στις υπηρεσίες. Έχουμε ήδη ξεκινήσει διαδικασίες παραβίασης κατά δύο κρατών μελών και έχουμε διάλογο με άλλα δύο, συγκεκριμένο διάλογο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε την όλη διαδικασία ώστε να εκμεταλλευτούμε απολύτως δυνατότητες που προσφέρει η οδηγία. Σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και αυτή είναι απλώς τεχνική διευκρίνηση, ε, για τα συστήματα επαγγελματικών συντάξεων θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι οι υπηρεσίες αυτές εμπίπτουν στη 2006-54 οδηγία, του ΡΙΚΑΣ δηλαδή, και έχουν χωριστεί αν θέλετε διακριτή εξέταση στο πλαίσιο αυτό. Εμείς έχουμε σημειώσει βεβαίως και την απόφαση τεστασσά και άλλη μια απόφαση ε, σχετικά με το σύστημα αυτό των συντάξεων προκειμένου να εξασφαλίσουμε απόλυτη συνέπεια στους διάφορους πυλώνες πρώτο, δεύτερο και τρίτο των συστημάτων συντάξεων. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Merci. Ευχαριστώ. Για την αλλαγή σκητάλης ε, χρειαστήκαμε κάποια δευτερόλεπτα. Ευχαριστούμε την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρία Ανίσκα Κοσλόσκα, η εισηγήτρια μήπως θέλει να δευτερολογήσει, να συνοψίσει οτιδήποτε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις παρεμβάσεις και τις παρατηρήσεις σας. Ε, είναι καυτό το ζήτημα και παρότι είναι Ιούλιος γίνεται αυτή η ζωηρή συζήτηση και σίγουρα με όλες αυτές τις παρεμβάσεις θα είναι πολύ καλή η τελική έκθεση. Ευχαριστούμε. θα την ε, ολοκληρώσουμε τώρα τη συζήτηση και θέλω μόνο να σας πω ότι οι δύο εμπειρογνώμονες θα μας στείλουν και επιπρόσθετες γραφές σε πληροφορίες, ε, γιατί υπάρχουν σίγουρα κάποια ζητήματα ε, για τα οποία μπορείτε να δώσετε και γραπτές απαντήσεις. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Θα περάσουμε στο επόμενο σημείο, αφού ολοκληρώσαμε τώρα αυτό το ζήτημα. Η συμβολή μας στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017. Κατά παράδοση, εκδίδει γνωμοδότηση η Επιτροπή μας. Η Σάνφρος Νταντζίλα είναι η συγγήτρια, αλλά επειδή απουσιάζει, θα ακούσουμε την κυρία Αρένα. Από την ίδια ομάδα είσαστε φυσικά. Άρα, να ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα πολύ γρήγορα να σας πω ότι η κυρία Ταντσίλα ε, ζητά συγγνώμη που δεν μπόρεσε να έρθει και θα σας διαβάσω εγώ τα σχόλιά της. Παρατηρεί η κυρία Τανσιλό ότι για να είναι ουσιαστική η πολιτική μας για των δύο φύλων θα πρέπει να ενσωματωθεί το θέμα και στις πιστώσεις, γραμμέ του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Εδώ στην Επιτροπή ζητάμε ξεκάθαρου δείκτες για την χρήση των πιστώσεων υπό αυτή την οπτική γωνία τη ισότητα των δύο φύλων και αυτό είναι σημαντικό για να γίνεται και αξιολόγηση. Η στρατηγική 2020 Επίσης πρέπει να προβλέπει τέτοιες πιστώσεις για την υλοποίηση αυτών των ειδικών στόχων, κυρίως σε προγράμματα όπως ε, Δάφνη, παραδείγματος χάρη κυρίως για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Πρέπει να ενισχυθούν αυτά τα προγράμματα. Ε, ποιες είναι οι τάσεις 2016-2017. Υπάρχει κάποια σταθερότητα σε σχέση με την πρικοδότηση του προγράμματος. Το 2011 είχε 20 εκατομμύρια ε, και τώρα δυστυχώς έχουμε πέσει στα 14,8. Ε, είναι λοιπόν σημαντικό να υπενθυμίσουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το πρόγραμμα για την καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Πρόεδρο. Εμεί σα ευχαριστούμε, κυρία Κοσλόσκα, για το ΕΛΚ, παρακαλώ. Θα ήθελα να ζη... Ε, ζητώ συγγνώμη εκ μέρου της κυρίας Ματέρα που απουσιάζει και θα ήθελα να διαβάσω ένα σημείωμα εξ ονοματό τη. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Τενσίλα για τη σημαντική δουλειά αυτή για το γενικό προϋπολογισμό του 2017. Το ΕΛΚ χαιρετίζει το κείμενο το οποίο είναι ισορροπημένο και συνεπές αλλά εκφράζουμε μία λύπη σχετικά με το πρόγραμμα Αντάφνε που δεν έχει πλέον γραμμή σχετικά με την καλύτερη προστασία των γυναικών, των παιδιών και των νέων στην Ευρώπη. Είμαστε υπέρ της ε, καλύτερης υποστήριξης των φορέων που επιτηρούν την ε, αποτροπή των διακρίσεων και της βίας κατά των γυναικών και συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες σχετικά με την επίτευξη των στόχων 2020 ε, του συνολικού επίπεδου απασχόλησης των γυναικών στο 75% και ότι περισσότερα πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης θα υποβάλουμε τροπολογίες για το γενικό κείμενο από την εμπειρία των τελευταίων ετών Στην Επιτροπή Προϋπολογισμού όμως ε, τα αιτήματα που προέρχονται από την Επιτροπή μας δεν είναι πολύ ψηλά στην ε, λίστα προτεραιοτήτων. Επομένως δεν πρέπει να ζητήσουμε και πάρα πολλά κατά την άποψή μας. Merci, Σας ευχαριστώ. Η κυρία Βανά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και στην εισηγήτρια για αυτήν την, ε, το εξαιρετικό σχέδιο γνωμοδότησης. Για μας είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και ακριβώς διότι συνδέεται με τον προϋπολογισμό ε, για ε, τα δύο φύλλα. Θεωρώ πως είναι πραγματικά ε, λυπηρό για το ότι δεν υπάρχει διοργανική συμφωνία για την κατάρτιση προϋπολογισμού ισότητας. Και θα υποβάλουμε σχετική τροπολογία έτσι ώστε να ζητήσουμε την Επιτροπή Γυναικό, από την Επιτροπή Γυναικών να συμπεριλάβει ε, το θέμα αυτό στον προϋπολογισμό. Επίσης, Στην γνωμοδότηση αναφέρονται μέτρα για την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας και το θεωρούμε ντροπή ε, ότι απέχουμε τόσο πολύ από τους στόχους του 2020 ε, για το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Θα υποφάλουμε λοιπόν ε, σχετικές τροπολογίες. Όπως επίσης και για την επενδυτική πολιτική και για το ότι πολλές γυναίκες ζουν στα όρια της φτώχειας. Θα υποβάλουμε επίσης τροπολογίες για την χρήση των διαρθρωτικών ταμείων και για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εδώ πιστεύω πως πρέπει να ενισχύσουμε ε, την συμμετοχή των γυναικών και επίσης θα, φέρουμε, θα υποβάλουμε μια τροπολογία για τις γυναίκες πρόσφυγες. Επιστώντας την προσοχή, την προσοχή στο ότι οι περισσότεροι πρόσφυγες είναι γυναίκες. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έχουμε κάποιον άλλο που θα επιθυμούσε να μιλήσει για, το... για τα θέματα προϋπολογισμού. Δεν βλέπω. Επομένως, να κλείσουμε και αυτή τη συζήτηση δίδοντας κάποια στοιχεία χροντιακράματος. Υποβολή τροπολογιών για την γνωμοδότηση της Επιτροπής ΦΑΜ θα κλείσει 15 Ιουλίου το μεσημέρι. οι τροπολογίες προϋπολογισμού μπορούν να εξακολουθήσουν με προθεσμία στις, μέχρι τις 23 Αυγούστου, μία η ώρα το μεσημέρι. Έχει προβλεφθεί να ψηφίσουμε επί της νομοδότησης της Επιτροπής μας στην συνεδρίασή μας μετά τις διακοπές 1η Σεπτεμβρίου. Αυτά επί του χρονοδιογράμματος για την γνωμοδότηση για τον προεκλογισμό 17. Και πάμε στο τελευταίο σημείο σήμερα, το οποίο μεταφέρθηκε από την εχθισινή ημερήσια διάταξη. Τα θεμελιώδη δικαιώματα και θα δώσω το λόγο στον κύριο Σεμπαστιά, τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη γιατί Είχα προβλήματα με την πτήση μου χθε. Άργησα δύο ώρες και δεν μπορούσα να φτάσω στην ώρα μου για την χθεσινή συνεδρίαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, ομάδα εργασίας, την γραμματεία, γιατί αντέδρασαν πάρα πολύ γρήγορα και κατάφεραν να αλλάξουν το ε, σημείο αυτό και να το μεταφέρουν σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Είναι μια πολύ σύντομη γνωμοδότηση. Ακριβώς επειδή μας περιορίζει ο χώρος, ο αριθμός των λέξεων, η γνωμοδότηση αφορά την, ε, την ισότητα των γυναικών. Θέλουμε να στείλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα ισχυρό μήνυμα ότι η ισότητα των φύλων είναι θεμελιώδες ε, στατικό στοιχείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο κείμενο πιστεύω υπάρχουν τρία διαφορετικά ε, θέματα. Τα αρνητικά σημεία όπου πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε απόλυτη ισότητα μεταξύ των δύο φίλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν είναι καθήκον μας να το αναφέρουμε ρητά. Έπειτα, υπάρχουν κάποια, κάποια αιτήματα. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη την εισαγωγή της συνεκτίμησης διάστασης του φύλου στην πολιτική της Ένωσης. Αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητούμε νομική πράξη, δεν διευκρινίζουμε τι, διότι αυτό είναι αποφάση της Επιτροπής, που να καταδικάζει την βία κατά των γυναικών. Θέλουμε ένα κοινό πλαίσιο ε, για να αντιμετωπίσουμε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το λόγο αυτό χρειάζονται καλύτερα δεδομένα, καλύτεροι δείκτες, Γι' αυτό λοιπόν στηρίζουμε την ε, δουλειά που κάνει το, ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ισότητας των Φύλων. Μετά ζητούμε από τα κράτη-μέλη την εφαρμογή ε, μέτρων όπου θα, ε, τα οποία θα προστατεύουν ε, τις ε, γυναίκες που ζητούν άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, κυρώσει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και Έχουμε ακούσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δύο φορές το έχουμε ακούσει αυτό, προτίθεται να κυρώσει τη σύμβαση φέτος. Εμείς ε, περιμένουμε λοιπόν αυτή την απόφαση, την καλωσορίζουμε και σε γενικές γραμμές αυτά περιέχει η γνωμοδότησή μας. Περιμένουμε τις τροπολογίες σας έτσι ώστε να βελτιώσουμε την γνωμοδότηση και να την ε, κάνουμε πιο ισχυρή. Θεωρώ όμως πως το μήνυμα είναι σαφές και πρέπει να, ε, ακολουθήσουμε, να επιμείνουμε διότι είναι καθήκον μας να προστατεύσουμε την ισότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Ας ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση. Ίσως οι σκιώδεις θα ήθελαν να μιλήσουν. Η κυρία Αγίνα. Μιλάω εξ ονόματος της κυρίας ε, Γιούτοβα που είναι υπεύθυνη για το φάκελο αυτό. Καταρχάς να συγχαρούμε τον ε, συνάδελφο τον κύριο Σεμπαστιά. Ε, συμφωνούμε απολύτως με την ανησυχίες που εκφράζει. Για μας το θέμα της ισότητας θα πρέπει να την χάνει οριζόντιας ε, χειρήσεως με ποσοτικοποιημένο τρόπο και να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι τομεί όπως και οι τακτικές αξιολογίες αντικτύπου που γίνονται στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 και μια ετήσια ανάλυση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που θα, έχουμε, θα μας επιτρέψει να έχουμε καλύτερη παρακολούθηση των πολιτικών. Και χθε ακριβώς το ίδιο προτείναμε προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη παρακολούθηση του αντικτύπου των πολιτικών που εφαρμόζονται. Ε, σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που έχει οδηγήσει σε ανεργία και επομένως και σε διακρίσεις, ιδιαίτερα κατά των γυναικών, η μεταναστευτική κρίση, η πολιτική κρίση ε, και η κρίση αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε όλο και πιο συντηρητικές απόψεις σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στην κοινωνία μας. Ε, τις περιορίζουμε στον πυλώνα, τον κοινωνικό και οικογενειακό, αθέλετε και ε, δεν τις συμπεριλαμβάνουμε στον, οικονομι... στον οικονομικό πυλώνα της κοινωνίας πλήρως. Εμείς δεν θέλουμε μια προσέγγιση σύμφωνα με την οποία κάποιο από τα δύο φύλλα θα έπρεπε να υπερισχύει σε οποιοδήποτε από αυτούς τους δύο πυλώνες. Θα πρέπει να έχουμε παρουσία και σε όλες αυτές τις περιοχές και σχετικά με τις ε, ε, άδειες μητρότητας αλλά και πατρότητος πρέπει να προσέξουμε σε όλα τα μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν την λήψη πολιτικών αποφάσεων και οικονομικών αποφάσεων εκ μέρους των γενικών και να καταπολεμήσουμε τα φαινόμενα βίας και ένα στοιχείο θα ήθελα να αναφέρω για τις οικογένειες μεταναστών ε, έχουμε μια πολύ μεγάλη, μεγάλη ποσόστοση ε, από τις μελέτες που δημοσιεύονται από τέτοιες οικογένειες παιδιών και γυναικών, επομένως πρέπει να το προσέξουμε. Σας ευχαριστώ. Για το ECR, κύριος Γκέρι, παρακαλώ. Yeah, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον συνάδελφο Σεμπαστιάν για την παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησης για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ε, μπορείτε να φανταστείτε, ε, εγώ προσωπικά αλλά και η ομάδα ECR δεν μπορούμε να ε, δεχτούμε και να συμφωνήσουμε με όλα τα σημεία. Καταρχάς, όσον αφορά το θέμα της ισότητας ως δείκτη για το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Ε, δεν συμμερίζομαι αυτήν την άποψη. Θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι ένα όργανο μέτρησης της οικονομικής ε, ε, δυνατότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι ως ένα συνονθήλευμα διαφόρων άλλων ενδείξεων. Έπειτα, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Σύμφωνα με τον ορισμό της Παγκόσμιας Διάσκεψης του 1994 στο Κάιρο για τον πληθυσμό αναφέρεται ότι ψυχική, σωματική και κοινωνική ε, υγεία συνδέονται άμεσα με την σεξουαλικότητα και την αναπαραγωγή. Εδώ θέλω να σας πω ότι πρέπει να κοιτάξουμε και ε, το, την πρόληψη των ε, αμβλώσεων κατά εξαναγκασμό και όχι να τις στηρίξουμε. Μετά, ε, χθες μιλήσαμε για έναν μισθό ανατροφής παιδιών. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί σε κανένα κράτος μέλος ακόμα. Οι γυναίκες είναι και μητέρες και θα πρέπει να έχουν ε, την ανεξαρτησία τους για να μπορούν να είναι μητέρες. Δεν θα πρέπει να αναγκάζονται να δίνουν τα παιδιά τους ε, σε άλλους για να τα μεγαλώσουν. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι ακριβώς και επειδή ένα παιδί μεγαλώνει καλύτερα μαζί με τη μητέρα μου πρέπει να υπάρχει δυνατότητα οι μητέρες ε, να στηρίζονται οικονομικά στην ανατροφή των παιδιών τους. Έπειτα, αυτό θεωρούμε είναι δημοκρατικό και πρέπει να υπάρχει σε ένα κράτος δικαίου. Σε γενικές γραμμές να πω ότι θα υποβάλουμε τις σχετικές τροπολογίες και παρότι δεν συμφωνούμε σε σημεία, ε, είναι γενικά καλή γνωμοδότηση. Ευχαριστώ κύριε Μπιόρκ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, θα μιλήσω στα αγγλικά. Θέλω να προσπαθήσω να επικοινωνήσω απευθείας μαζί σας. Συμφωνούμε ε, σε πολλά πράγματα. Ξέρω ότι είσαστε φεμινιστής όπως και εγώ. Είμαι φεμινίστρια. Ε, για δικαιώματα ΛΟΑΤ και ούτω καθεξής θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες. Ελπίζω να τις συνυπογράψουμε. Έχω και άλλα ζητήματα που έθεσε και, έθεσαν και οι σοσιαλιστές ε, για το αντιφεμινιστικό και αντιλόατ κίνημα σε κάποιες χώρες που απειλεί τα δικαιώματα των γυναίκων. Επίσης ε, για τις αιτούσες άσυλο θέλω να ενισχυθούν τα δικαιώματά τους, το ίδιο και για την οικογενειακή επανένωση, διότι έτσι παραβιάζονται κυρίως δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών. Οι ΡΟΜ γυναίκες ε, είναι μια ομάδα που εξακολουθεί να είναι πολύ εκτεθειμένη, παραβιάζονται κατάφορα τα ε, δικαιώματά τους. Θα καταθέσω σχετικές τροπολογίες και μετά... επειδή ασχολούμαστε με τα δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, ούτως ή άλλως εδώ στην Επιτροπή Γυναικών, θα καταθέσω ε, κάποιες τροπολογίες ε, για το δικαίωμα στην άμβλωση, στην σεξουαλική κατάρτιση ε, είναι βασικά δικαιώματα στην Ευρώπη. Και υπάρχουν και κάτι άλλα, Τζόρντι, κάποια άλλα στήματα που ίσως δεν μας βρίσκουν σύμφωνος. Περιμένω, περιμένω. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, αλλά εγώ, ε, όταν θεωρώ ότι πρόκειται για βασικά δικαιώματα των γυναικών για το σώμα τους, για τη σεξουαλική τους υγεία και μιλώ εδώ για τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την πορνεία, δεν μιλάω για συντηρητισμό ή για ε, ηθικολογική προσέγγιση. Το αντίθετο είναι. Ε, μέσα σε αυτές τις αγορές πορνείας ε, δεν υπάρχει τίποτα πιο συντηρητικό γιατί ε, ο έλεγχος ε, σεξουαλική των σωμάτων των γυναικών, η σεξουαλική τους εκμετάλλευση είναι το αντίθετο. Το ίδιο για την παρένθετική Νομίζω ότι ε, αγοράζουμε και πουλούμε τα σώματα των γυναικών ε, σε, με τρόπο που ε, τις, ε, που έχει το αποτέλεσμα να περιέρχονται σε πάρα πολύ ευάλωτη θέση και γι' αυτό θα ήθελα από αυτή την πλευρά να μιλήσω για τις δομές εξουσίας και να προβάλλουμε τα δικαιώματα των γυναικών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα την κατανόησή σας ώστε ε, να πω και εγώ δύο λόγια γιατί αντικαθιστώ την ε, κυρία Πετή την σκιώδη του ΕΛΚΑ που δεν μπορέσει να παρακολουθεί στην αλλαγή ωραρίου και μου ζήτησε να διαβάσω ένα σημείωμα που είχε προετοιμάσει και το είχε προετοιμάσει στα αγγλικά. Άρα λοιπόν θα μιλήσω στα αγγλικά εκ μέρους της κυρίας Πετή η οποία λοιπόν ευχαριστεί ε, τον ε, κύριο Σεμπαστιά για το σχέδιο αυτό Θα ήθελε όμως εκ μέρους του ΕΛΚ να πει η κυρία ε, Πετή ότι δεν είναι 100% ικανοποιημένη από το σχέδιο αυτό και βλέπει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Κατά την άποψή της δεν καλύπτονται όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και όλα τα δικαιώματα τους που παραβιάζονται. Ε, θεωρεί ότι το κείμενο τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο δεν καλύπτει τις διακρίσεις κατά των γυναικών στον κόσμο των επιχειρήσεων και της επιστήμης ή των διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες στην ύπεθρο. Επίσης δεν βλέπει να γίνεται ιδιαίτερη μνήμα ε, στις διακρίσεις ή στο χώρο εργασίας κατά των γυναικών. Και δεν λαμβάνει υπόψη το σχέδιο ότι οι γυναίκες πλήττονται κυρίως από την ίνδια. Και υπάρχουν πολλαπλές μορφές και πολλαπλά επίπεδα διακρίσεων Επίσης υπάρχουν αυξανόμενα φαινόμενα βίας ε, κατά των γυναικών ε, ε, στο διαδίκτυο, στο οποίο επίσης δεν γίνεται αναφορά, ή στην εμπορία ανθρώπων και ιδιαίτερα γυναικών και νεαρών κοριτσιών. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα έπρεπε το σχέδιο αυτό να συμπληρωθεί και να ενισχυθεί ώστε να αποτελέσει μια πολύτιμη ε, ε, συνεισφορά. Η παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν θα πρέπει να αναφέρεται με τρόπο επιφανειακό. Θα πρέπει να δίδεται σε τέτοια κρούσματα επαρκής προσοχή. Εκ μέρους λοιπόν του ΕΛΚ θα υποβληθούν κάποιες τροπολογίες προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του σχεδίου και της συμπλήρωσης του σχεδίου. Επί τη βάση συγκεκριμένων και αυτών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και που δεν αναφέρει το σχέδιο. Και μία λέξη που θα ήθελε να αναφέρει η κυρία πετύχει για την προθεσμία των τροπολογιών. Ότι σε, αυτό σε αυτή τη φάση είναι αρκετά ασθενές οι προθεσμίες. Υποτίθεται ότι πρέπει να υποβληθούν όλες οι τροπολογίες μέχρι τις 18 και να ψηφίσουμε στην Επιτροπή Γυναικών 1η Σεπτεμβρίου και ως κοιόδη συγκήτρια έχει να πει η κυρία αυτή ότι καθότι η ψήφος στη Λίμπε έχει προγραμματιστεί στις, για τις 18 Νοεμβρίου αν ακούσαμε καλά την ομιλήτρια υπάρχει περιθώριο να αναβληθεί ο ψήφος, η ψήφος ε, στην Επιτροπή αυτή. Δεδομένης της διαφοράς, της απόστασης μεταξύ των δύο ημερομηνιών, ώστε να καταβάλουμε μια συλλογική προσπάθεια ε, προκειμένου να βελτιωθεί το κείμενο. Θα ζητήσουμε λοιπόν αναβολή της ψηφοφορίας διότι θεωρούμε ότι ε, το περνάμε λίγο στα γρήγορα το κείμενο, την όλη διαδικασία και δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Αυτό ήταν το τελευταίο σημείο που ήθελε να υπογραμμίσει εκ μέρους του ΕΛΚ και επανέρχομαι στη μητρική μου λέει πλέον η Πρόεδρος ζητώντας την κατανόησή σας. Νομίζω ότι κάποιοι έχουν ζητήσει το λόγο, η Κομισιόν καταρχάς. Παρακαλώ. Thank you, Madam Chair. Um... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Θα θέλαμε να κάνουμε ένα μόνο σχόλιο σχετικά με την πρόταση παριθμών 5, μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία των γυναικών μεταναστών και τον άσυλο. Αύριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τη νέα πρόταση για το άσυλο, η οποία περιλαμβάνει ε, διαδικαστικές δικλίδες, ιδιαίτερα για ε, τούντες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, γυναίκες και παιδιά για παράδειγμα. Αυτό που λάβαμε ιδιαίτερα υπόψη είναι οι ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών που ζητούν άσυλο οι οποίες ε, υφίστανται έμφυλη βία. Ε, πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, ε, συμβουλευτική ε, ψυχολόγων και όπως ε, και πριν, το ε, συμφέρον του παιδιού είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας. Υπάρχουν αρκετά μέτρα τα οποία ε, προτείνουμε για να διασφαλίσουμε την σωστή και ασφαλή κυδαιμονία των ασυνόδευτων ανηλίκων. Σας ευχαριστώ. Ναι, να ξαναδώσουμε το λόγο στον κύριο Σεμπαστιά για την τελευταία λέξη εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις προτάσεις σας. Καταρχάς συμφωνώ με όλους. Η γνωμοδότηση είναι πολύ σύντομη και δεν αρκεί ο χώρος που έχουμε για να, να ασχοληθούμε με ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ε, γι' αυτό λοιπόν ελπίζω οι τροπολογίες σας να βελτιώσουν το σχέδιο γνωμοδότησης έτσι ώστε να το κάνουν πιο πλήρες. Άκουσα πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις και θα ήθελα να τις συμπεριλάβω στη γνωμοδότηση τους σοσιαλδημοκράτες νομίζω αναφέρθηκε η διάσταση της οικονομικής κρίσης. Μετά. Το ΕΛΚ έκανε μια πρόταση σχετικά με την ε, διάκριση βάρος των γυναικών επιχειρηματιών, κάτι το οποίο φυσικά και πρέπει να συμπεριλάβουμε στη γνωμοδότηση. Οι γυναίκες επίσης είναι ε, θύματα διακρίσεων, θύματα φτώχειας, κινδυνεύουν περισσότερο να πέσουν ε, κάτω από τα όρια της φτώχειας από ότι οι άντρες και αυτό μπορούμε να το συμπεριλάβουμε στη γνωμοδότηση. Επίσης, εκπρόσωπος της Γκουε νομίζω μας είπε ε, για την επανένωση οικογενειών στην περίπτωση μεταναστών και όσον αφορά τις γυναίκες Ρώμα να μην ξεχνάμε ότι είναι η πιο ευάλωτη ομάδα γυναικών στην Ευρώπη και ε, θα ήθελα να συμπεριληφθεί και αυτό στη γνωμοδότηση. Τώρα, η πορνεία ως σεξουαλική εκμετάλλευση, αυτό είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα. Εγώ προσωπικά συμφωνώ απόλυτα με την άποψή σας, κυρία Μπιόρκ. Ε, τώρα, η θέση της ομάδας ECR. Θεωρώ καταρχάς πως πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και να ζητήσουμε να συμπεριληφθεί η συνεκτίμηση της διάστασης του φίλου στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Είναι σαφές από όλες τις συνθήκες ότι αυτό καθιστά προτεραιότητα και πρέπει να ζητήσουμε κάτι τέτοιο ακριβώς γιατί είμαστε και Επιτροπή Γυναικών. Στο θέμα των αυλώσεων τώρα θα ήθελα να σχολιάσω ότι αυτό συμπεριλαμβάνεται σε ένα σημείο που αναφέρει ότι ε, πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των γυναικών μεταναστών. Οι περισσότερες, αν όχι όλες, γυναίκες μετανάστες είναι θύματα βιασμού. Αυτό αναφέρεται ε, σε ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τι γίνεται όμως αν μετά από ένα βιασμό μια γυναίκα μείνει έγκυος. Εδώ ε, στεκόμαστε κι εμείς για το δικαίωμα των αμβλώσεων στις ε, γυναίκες. Πρέπει να σεβόμαστε τα δικαιώματά τους. Ξέρω πως είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα, αλλά πρέπει να σεβόμαστε τα δικαιώματα των γυναικών. Γι' αυτό λοιπόν και, χρησιμοποίησαμε την γνωμοδότηση για να εισαγάγουμε αυτό το σημείο, διότι θεωρούμε πως ε, αξίζουν σεβασμό γυναίκες και πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν τι θα κάνουν με το σώμα τους. Αυτά λοιπόν, περιμένω τις τροπολογίες σας. Και κάτι τελευταίο, ε, ψηφοφορίες. Δεν ξέρω αν μπορούμε να καθυστερήσουμε την ψηφοφορία, διότι η ψηφοφορία προβλέπεται για αρχές Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή. Δεν νομίζω λοιπόν πως είναι δυνατόν να αλλάξουμε κάτι στην μέση διάταξη. Δεν ξέρω, κυρία Πρόεδρε, ίσως έχετε κάτι να πείτε ή να προτείνω στη γραμματεία να εγώ να αλλάξουμε την ψηφοφορία. Ξέρω όμως ότι δεν είναι εύκολο. Γιατί υπάρχει θέμα χρόνου. Ωραία, ευχαριστώ. Συνάδελφε. Για το χρονοδιάγραμμα επαναλαμβάνω κάποια πράγματα για την υποβολή τροπολογιών. Επιβαίνω τη ημερομηνία ε, το 18 Ιουνίου μέχρι τις 6, ε, Ιουλίου, συγγνώμη, μέχρι τις 6. μετά από τι καρποφόρε συζητήσει του εισηγητή με του κοιόδε εισηγητέ, ενδεχομένω να υπάρξουν τροποποιήσει. Προ το παρόν πάντως προβλέπεται ότι την 1η Σεπτεμβρίου, την πρώτη συνεδρία μετά το καλοκαίρι δηλαδή, θα το συζητήσουμε και μετά 10 ε, και 11 Οκτωβρίου είναι, υπάρχει και άλλη συνεδρίαση της Επιτροπής Γυναικών. Θα δούμε αν θα αναβληθεί το ζήτημα. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε σήμερα γιατί θα το συζητήσουν οι συντονιστές και θα πρέπει να ε, καταλήξετε σε συνεννόηση. Επισήμως πάντως η ψηφοφορία έχει προβλεφθεί για την πρώτη συνεδρία, 1η Σεπτεμβρίου. Α, ναι. 31 ε, ε, Αυγούστου δεν συνεδριάζουμε, το επαναλαμβάνω όπως αρχικά έχει προβληθεί, δεν θα υπάρχει συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση στο το καλοκαίρι είναι σε 9 1η Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα το πρωί. Και εφόσον ολοκληρώσαμε την ημερήσια διάταξη, τη χτεσνή και τη σημερινή, καλό οι καλές διακοπές ευχαριστώ τη Γραμματεία της Επιτροπής, ε, το προσωπικό των ε, πολιτικών ομάδων, τους βοηθούς, ε, η, πρόεδρος, η Προεδρεύουσα ευχαριστεί και τους δημιουργούς, ευχαριστούμε και εμείς. Καλό καλοκαίρι.